Liebe Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάτσετε στις θέσεις σας like to proceed to the votes. για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Yeah. Liebe Kollegen, darf Sie herzlich begrüßen. Θα ήθελα να σας ε, ε, Καλώ ορίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, στη σημερινή μα συνεδρίαση. Καταρχήν, έχουμε την ψηφοφορία τη προσωρινή έκθεση, όπω ξέρετε. που εξετάστηκε στην Επιτροπή μα την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, την Πέμπτη στο Στρασβούργο και μετά τις ψηφοφορία έχουμε μια συνάντηση των συντονιστών για να αλλάξουμε τι ε, απόψεις μας όσον αφορά τη μελλοντική εργασία τη επιτροπή μα. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτο σημείο ψηφοφορία. Δεν υπάρχει τίποτα το ειδικό σαν πληροφορία, δήλωση κλπ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε μέσα στο σημείο 3 της σημερισίας μας διάταξης. Και ήθελα να τονίσω ότι είναι σύμφωνο με το καταστατικό μας να ψηφίσουμε σήμερα. Εξετάστηκε αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ψηφίσουμε πάνω στη συμβαστική αυτή πρόταση. Θα ήθελα να πω ότι άμα ψηφίσουμε πάνω στη συμβαστική αυτή πρόταση, αυτό σημαίνει ότι η αρχική έκθεση της Περβάνς Περές και οι 1625 τροπολογίες θα είναι πια χωρίς αντικείμενο. Äh, Μάρτιν. αναφερώ στη συμβαστική πρόταση, Πρόεδρε σαν ανεξάρτητο μέλος του Κοινοβουλίου εδώ, ότι δεν ανήκω δηλαδή σε κανένα κόμμα, δεν μπόρεσε το δικό μου γραφείο να πάρει ποτέ το... κοινοβούλιο. Διστάσαμε πολύ, υπήρξε βεβαιότητα για το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να κινητοποιηθεί και να κινητοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, τα, τους άσους που έχει στο μανίκι της, για να βοηθήσει τους πολίτες και να φανεί αυτό ολόκληρο τον κόσμο. Οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, τελικά, με την θέληση όλων των μελών της Επιτροπής αυτής, είναι κάτι που πιστεύω δείχνει και πόσο καλά εσείς προεδρεύσατε των εργασιών αυτών. Δείχνει επίσης πως όλοι βάλαν ε, ο καθένας το δικό του πετραδάκι για να καταλήξουμε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Κοιτώντα τώρα το περιεχόμενο του κειμένου, εννοείται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από το σημείο κίνησης μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Όμως πιστεύω ότι κάθε πρόταση είναι μια δυνατή πρόταση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να κάνει. Έπρεπε για να ακουστεί αυτό στα κράτη-μέλη, να ακουστεί στα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά για να το ακούσουν και οι πολίτες μας. Αποτελεί ένα βήμα, ένα στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Πρέπει να κινητοποιηθούμε ώστε η ψηφοφορία στην Ολομέλεια να δείξει ότι υπάρχει ο ίδιος δυναμισμός και σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο όπως υπάρχει σε αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μερικές φορές χρησιμοποίησαμε πλάγιους δρόμους, μερικές φορές ε, ε, καινοτομήσαμε. Αποφύγαμε κλασικές μεθόδους κοινοβουλευτικών εργασιών. Μετά, στη συνέχεια, θα πρέπει ο καθένας από εμά να μεταφέρει το μήνυμα αυτό πιο έξω, ώστε το μήνυμα αυτό να αποτελέσει και τη βάση της θέλησής μας για να παρέμβουμε και να επηρεάσουμε την πορεία των πραγμάτων. Αυτό περιμένει ο κόσμος από εμά. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, Είμαστε αποφασισμένοι μέσα στην ομίχλη που επικρατεί στην Ευρώπη, μέσα στην αβεβαιότητα αυτή που επικρατεί για πολλά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες μας. Εμείς λοιπόν θέλαμε να αποτελέσουμε το χώρο εκείνων όπου να μπορούν να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Αυτό το οποίο θετήσαμε, το κείμενο αυτό, αποτελεί πιστεύω μια πολύ καλή βάση για να γίνει, για να δώσουμε τον αγώνα αυτόν απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέρφους για την αποφασιστικότητα που δείξανε, για τη θέλησή τους και μαζί σας μοιράζομαι τη χαρά μου για ένα κείμενο το οποίο πιστεύω δίνει το μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα στην Ευρώπη και ότι εξαρτάται από τη δικιά μας αποφασιστικότητα, από τη δικιά μας την βούληση να ε, αντιδράσουμε και να καταπολεμήσουμε τις αδράνειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Περβάτσο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτό. Όσον αφορά την χρονική οργάνωση, δεν μπορούσαμε καλύτερα να ψηφίσουμε παρά σήμερα γιατί αυτή την εβδομάδα θα υπάρχουν προτάσεις του Πρόεδρου ε, Φανρόπρε, της Εκτελεστικής Επιτροπής επίσης. Το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα και είναι πάρα πολύ καλό και σημαντικό να ακουστεί σε αυτό το θέμα και η φωνή του Κοινοβουλίου. Και ότι εκφραζόμαστε με μεγάλη πλειοψηφία, παρόλο που πολιτικά βέβαια οι απόψεις μας σε πολλά σημεία απέχουν, δείχνει ότι πραγματικά και το Κοινοβούλιο σε περίοδους κρίσης μπορεί να μιλήσει με μία φωνή. Ευχαριστώ όλους που συνεργάστηκαν εδώ. Ολοκληρώνεται εδώ η ψηφοφορία. Παρακαλώ τώρα τους συντονιστές να παραμείνουν στη αίθουσα γιατί έχουμε τώρα μια συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.